εδάφιο ε, 6 του κανονισμού ενημερωνόμαστε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από τη διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στην σύσταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων να μην αντιταχθεί σε κατεξιζόδοτηση πράξη. Εάν εντός 24 ωρών καμία πολιτική ομάδα ή αριθμός μελών που να είναι, ίδιο, ε, που να είναι ίσο με το ελάχιστο όριο δεν εκφράσουν αντιρρήσεις, η σύσταση αυτή θα θεωρηθεί εγκεκριμένη. δάλος θα ψηφιστεί. Η ε, σύσταση αυτή διατίθεται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας.